στην ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ε, γιατί φυλακίσατε τους καταλανούς ηγέτες πέρσι. Πιο καλά στην Τουρκία είμαστε, στην Ισπανία και όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έπρεπε να γίνει ρεφερέντουμ, δημοψήφισμα που δεν είναι έγκλημα για τη μεταρρύθμιση του Θαπατέρωτο από το 2005. Επίσης, κανονικά ε, υποτίθεται ότι τα καταλανικά είναι επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο φετεραλισμός είναι να μπορούμε να μιλάμε τη γλώσσα του άλλου. Ποια μέρα θα μιλήσουμε καταλανικά εδώ μέσα και έπειτα. Στην Καταλωνία δεν έχουμε πρόβλημα συμβίωσης. Το πρόβλημα είναι η κεντρική κυβέρνηση της Ισπανίας. Στο διάλογο θα τα βρούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. μου κύριε Πρόεδρε να ξεκινήσω λέγοντας ε, ότι ε, αφού αναφέρεστε για τον εξτρεμισμό το πρόβλημα είναι ότι στην πραγματικότητα δεν ε, εφαρμόζεται τίποτα από τις αρχές σας. Αυτή τη στιγμή ε, μια πρόταση εμπιστοσύνης τελικά τερμάτισε τη θητεία του Ραχώη. Εσείς πέσατε στην αγκαλιά των πολιτικών κομμάτων των ε, αποσχιστών οι οποίοι προσπάθησαν να διαρρήξουν τη συνταγματική τάξη, οι οποίοι παρεκτράπηκαν από τον νόμο και δεν έχουν καμία δημοκρατική νομιμότητα. Κύριε Πρωθυπουργέ, μπορείτε να έρθετε εδώ και να μας αφήσετε μια ιστορία, αλλά όταν στο τέλος η πραγματικότητα και τα δεδομένα τελικά αποκλίνουν τόσο πολύ, θα συνειδητοποιήσετε τι γίνεται. Πρέπει να υπάρχει συνέπεια και εσείς δεν έχετε καμία απολύτως συνέπεια και το αποδείξατε. Mr. Prime Minister κύριε Πρωθυπουργέ, Αναφερθήκατε στη νέα νομιμοποίηση της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Ζητήσατε περισσότερη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Δεν πιστεύετε ότι οι πολίτες ε, βρίσκουν ότι έχουν στερηθεί την κυριαρχία τους, ε, δεν μπορούν πια να αποφασίσουν για το ίδιο το μέλλον τους. Βλέπουμε από βιομηχανοποίηση ε, και εγκατάλειψη πολλών περιοχών και οι άνθρωποι που μένουν εκεί ε, θεωρούν ότι δεν έχουν ελέγγυν ως προς το πώς ε, θα εξελιχθεί η ζωή τους. Πώς βλέπετε εσείς την κυρίαρχη δημοκρατία η οποία με νέο τρόπο θα αντιστοιχεί στην επιθυμία των πολιτών να έχουν λέγει όσον αφορά το μέλλον τους. Όλα αυτά ε, σε συνδυασμό με την ιδέα ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα νέο ξεκίνημα. Αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ, ήταν κεντρικό σε όλα τα θέματα που συζητήθηκαν από το Brexit μέχρι την Καταλωνία. Ευχαριστώ, Σαλαφράγκα. Πρόεδρε, Κύριε Πρόεδρε τη Κυβέρνηση, καλώ ορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το είπατε με βεβαιότητα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε αξίε. Γι' αυτό αυτό το Κοινοβούλιο έχει ε, ε, μια παρέγκλητη δέσμευση με τα ανθρώπινα δικαιώματα σε οποιαδήποτε χώρα ή ήπειρο. Ε, είναι καθολικά τα ανθρώπινα δικαιώματα, γι' αυτό και φτιάξαμε αυτό το βραβείο για την ελεύθερη ε, συνείδηση που ονομάζεται Ζαχάροφ. Εγκρίναμε τρία, έχουμε δώσει μάλλον ε, στον Οσβέλτο Βάνια, τον Γουλιέλμο Φαρίνια και πέρσι στην Δημοκρατική Αντιπολίτευση της Βελεζουέλας ε, τα βραβεία Ζαχάροφ. Εσείς τι άποψη έχετε. Πιστεύετε ότι οι βραβευμένοι είναι αξιόλογα άνθρωπα, τα ε, άτομα τα οποία υπερασπίζουν την ελευθερία και την αξιοπρέπειά τους, είτε είναι στην Κούβα είτε είναι στη Βενεζουέλα. Θα είσαστε διαθέσιμος να συναντηθείτε μαζί του και σε σχέση με τη Βενεζουέλα έχουμε ε, με μεγάλη πλειοψηφία ψηφίσει ψήφισμα που ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να ε, ζητήσουν ε, ε, να γίνει έρευνα από το, Ευρωπα... από το Διεθνές Δικαστήριο για τα εγκλήματα που έχουν γίνει σε αυτή τη χώρα. Και ποια είναι η γνώμη σας αν ζητήσουμε από τον Καναδά και τις είπα να συμφωνήσουν για αυτή τη διαδικασία. Κυρία Βαλενσιάνο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, εσείς σκεφτήκατε ότι το ο ΕΛΚ ε, που έχασε την πλειοψηφία. Όχι. Ε, το ΕΛΚ ζητάει ένα πατριωτισμό όταν είναι στην αντιπολίτευση αλλά οι ίδιοι από την πλευρά τους δεν ε, το κάνουν όταν εμείς είμαστε στην κυβέρνηση. Η βασική ιδέα που διαβιβάσατε εδώ είναι ότι πνέει ένας αέρας λαϊκισμού ε, κατάτμισης, διέρεσης εξτρεμισμού στην Ευρώπη, ε, αντιδραστικού πνεύματος έναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έναντι στην ισχύ της Ένωσης, έναντι στην ε, ισχύ των γυναικών. Πρόκειται για μια, ένα αντιδραστικό λαϊκιστικό κίνημα που λέει ότι δεν έχει συμπλέγματα, αλλά ούτε εμείς έχουμε συμπλέγματα. να πάμε μπροστά φιλοευρωπαϊστές χωρίς συμπλέγματα.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 Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπνευσμένη ομιλία σας για την Ευρώπη των ανθρώπων, μια ομιλία που δίνει ελπίδα και θάρρος. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τις γυναίκες. Έχουμε διαπραγματευτεί στο Κοινοβούλιο εδώ και πολύ καιρό μια έκθεση που προβλέπει οι άντρες και οι γυναίκες να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στα διευθυντικά συμβούλια επιχειρήσεων. Εσείς ε, μιλήσατε υπέρ της ιδέας αυτής και ε, απευθύνομαι και στον ε, Πρόεδρο Ταγιάννη. Κατά τον χρόνο ομιλίας φροντίζεται εξίσου να μιλούν οι γυναίκες ώστε να μην έχουμε ανισορροπία διότι για να λύσουμε το θέμα της ισότητας θα πρέπει να ακούγεται περισσότερο και η φωνή των γυναικών στο Κοινοβούλιο. Ε, Σα θυμίζω ότι είναι κάποιοι που έχουν υπογράψει την πρόταση τη. Κομισιόν. Ε, είμαι ένα από αυτού που έχουν υπογράψει την πρόταση τη Κομισιόν για περισσότερε ε, θέσει για τι γυναίκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το λόγο έχει η κυρία Κοράτσα Μπίλτε. Κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ. Κύριε Πρωθυπουργέ, συμμερίζομαι τις ανησυχίες σας για την αντιευρωπαϊκή ρητορική από την ακροδεξιά και την ανάγκη για ανανέωση της νομοποίησης ε, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Το Κοινοβούλιο πάντα ψηφίζει ξεπερνώντας τα ε, κομματικά και εθνικά όρια για ενιαία έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλουμε εμείς να αποφασίζουμε που θα συναντιόμαστε και που θα συζητάμε. Και η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Κούρτς μίλησαν υπέρ της μίας έδρας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εσείς ως ε, φιλοευρωπαίος ε, είσαστε διατεθμένοι να στο Συμβούλιο και κατά το προεκλογικό αγώνα να μιλήσετε στους ανθρώπους της Ισπανίας και της Ευρώπης ε, για το θέμα αυτό ή θα αγνοήσετε το θέμα αυτό και θα διακινδυνεύσετε ένα σύμβολο Ευρώπης και συμφιλίωσης στην Ευρώπη, κάτι τόσο αγαπητό σε όλους εμάς, να γίνει ε, σύμβολο σπατάλης. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Revolta Land Bonfoy. Αγαπητέ Πρωθυπουργέ, σα ευχαριστώ για την ομιλία που κάνατε. Ευχαριστώ για αυτή την ομιλία που μας δίνει ελπίδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί προτάσει τα κοινωνικά, οικολογικά ε, θέματα, τα θέματα αλληλεγγύη και αξιών και τα ε, θέματα του Ευρωπαϊκού ε, Προπολογισμού. Εκφράσατε μεγάλες φιλοδοξίες λέγοντα ότι το 1% του ΑΕΠ των κρατών μελών δεν αρκεί για να έχουμε ισχυρές ευρωπαϊκές προτάσεις. Επίσης, τολμήσατε να μιλήσετε για Ομοσπονδιακή Ευρώπη και αυτό πολύ μα χαροποίησε. Σα ευχαριστώ γι' αυτό. Να επανέλθω στην κατάσταση στην Ανταλουσία. Ανησυχούμε πάρα πολύ εδώ και χρειαζόμαστε οπωσδήποτε να σταματήσουμε κάθε είδους αμφισημία ή παραφύση συμφωνίας ανάμεσα σε, αρχές της σε δυνάμεις της δεξιάς και της ακροδεξιάς. Είναι σημαντικό να τονίζουμε αυτή τη συμμαχία και την προοδευτική αυτή ε, συμμαχία. η τώρα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα διαδικαστικό. Καταρχάς θέλω να απορρίψω και να εκφράσω τη λύπη μου που επιτρέπετε να βάλετε, ε, ε, να, να, να, να αναρτώνται εδώ αφήσει από ε, κρατούμενους. Είναι έλλειψη συμβασμού στον πρόεδρο της κυβέρνησης της Ισπανίας αυτό. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Κύριε Σάντσες. Εσείς ήρθατε ζητώντας να προστατευτεί το ευρωπαϊκό μοντέλο και κάποια άλλα πράγματα από τους ακραίους που το απειλούν. Μπορώ να σας πω ότι ε, εσείς μιλάτε για τους ε, εξεμισμούς στην Ευρώπη, αλλά παρακαλώ εξηγήστε μας και σε ολόκληρη την Ευρώπη ότι εσείς είστε πρόεδρος της κυβέρνησης Ισπανίας ακριβώς χάρη σε αυτούς τους εξεμιστές. Δηλαδή, στο του της Καταλωνίας από το Χάριστο στο του που πάει χέρι-χέρι με τους τρομοκράτες του ΕΤΑ που εντάξει κάποιες φορές ε, ε, έκαναν και πολύ ντροπιαστικά θέματα. Κύριε Σάντσες, πώς μας να μας εξηγήσετε με, ότι συγκυβερνάτε με αυτούς που είναι οι μεγαλύτεροι απαταιώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής. Ευχαριστώ. Λόπες, Χάβι Λόπες. Βρε κύριε Ε, φέρατε εδώ τη φωνή των φιλοευρωπαϊστών υπέρ μιας κοινωνικής Ευρώπης που φροντίζει την ε, επισφάλεια των θέσεων εργασίας κλπ. Μια Ευρώπη οικολογική η οποία ηθήνεται του αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Μια ανοιχτή Ευρώπη η οποία θεωρεί ότι η ανοχή και απέναντι στον άλλον είναι λόγος ε, ύπαρξης. Μια Ευρώπη φεμινιστική που θεωρεί την ισότητα των φύλων έμβλημά τη. Αυτή είναι η φωνή της Ισπανίας σήμερα. Μια φωνή που χρειαζόμαστε οι Ευρωπαίοι και που γίνεται καλώ δεκτή από αυτό το σώμα. Μια Ευρώπη η οποία κατανοεί ότι το μέλλον της θα περάσει μέσα από την ε, ε, οικοδόμηση μια κοινή ε, ηθαγένεια και μετατρέπει τον διάλογο και την συμβίωση σε λόγο ύπαρξή της. Επίσης στην Καταλωνία προσπαθείτε να ξεκινήσετε τον ε, διάλογο ε, ε, επιστρέφοντας πολιτικές λύσεις. Αυτή είναι η μόνη λύση για το μέλλον των Καταλανών, ο διάλογος. Ο κύριος Σωμάτο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Σάντσεθ, ε, περίμενα τουλάχιστον ε, σε μια μιλία που διέρχεται 37 λεπτά να αφιερώσετε 10 δευτερόλεπτα να αναφερθείτε για παράδειγμα στα Κανάρια. Μιλάτε για, τα, για το μέλλον της Ευρώπης αλλά περνάει και από, αυτή την, και από αυτές τις απομακρυσμένες περιφέρειες που χρήζουν στήριξης. Ε, οι Κανάριοι νήσοι ε, έχουν γίνει τουριστικός προορισμός. Ε, Παρ' όλα αυτά θα έπρεπε να είναι κάτι παραπάνω, ένα υπόδειγμα της πολιτικής συνοχής και πολιτικής αλληλεγγύης. Ο κύριος Ταχάνη τόνισε τη σημασία του και είναι αλήθεια. Εμπιστεύομαι ότι ε, θα αποκτήσει και για σας ε, αυτή τη σπουδαιότητα να εκπληρώσετε, να εφαρμόσετε τις ε, συνθήκες, συμφωνίες με τις περιφέρειες αυτές και να τους δείξετε ότι από εδώ, από την καρδιά της Ευρώπης θα έχουν την, υποστήριξη, την πλήρη μας υποστήριξη. Κύριε ευχαριστώ. Ε, στην κυβέρνησή σας και στον Υπουργό Εξωτερικών σας, Γιουζεφ Μπορέλ, που ήταν πρώην Πρόεδρος αυτού του Κοινοβουλίου. Θέλω να τονίσω από την ομιλία σας τη λέξη φεδεραλισμός. Η ανάγκη να εξακολουθήσουμε να ζητάμε την οικοδόμηση μιας ομοσπονδιακής Ευρώπης, που είναι μια ιδέα για την αναδιοργάνωση και της χώρας μας της Ισπανίας, που δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά την αναγνώριση της αρμονίας και την δυνατότητα να ζήσουμε με ελευθερία και ειρήνη. Χρειάζεται αυτό για να προστατεύσουμε την Ένωση και τους πολίτες. Αρμονία που τη χρειαζόμαστε για να προστατεύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση που χρειάζεται να μεταρρυθμιστεί, να μεταρρυθμίσει της Νομισματικής Ένωσης. Χρειάζεται και ο φορολογικός πυλώνας για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια για την ανεργία. Πρέπει να φτιάξουμε μια πλειοψηφία για τις πρόκειτες προς... επόμενες εκλογές με την Κομισιόν ε, για να έχουμε μια ασφάλιση για την ανεργία που να προστατεύει τους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος ο κύριος Μίγιαν Από την ένταξη της Ισπανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το θέμα της, ε, ε, των σχέσεων της Ισπανίας με τη Λατινική Αμερική ήταν σημαντικό για κάθε Ισπανό ηγέτη. Πώ σήμερα αποφύγατε να αναφέρετε όχι μόνο τη Βενεζουέλα, αλλά και τις πολύ σημαντικέ προματεύσει με το Μερκοσούρ, κύριε Πρόεδρε, στην ομιλία σας. Μ' ανησυχεί αυτό που είπατε, ανησυχούν αυτό που είπατε, αλλά και αυτά που δεν είπατε. Κάτι ακόμα που θέλω να τονίσω είναι το Brexit και συγκεκριμένα τα θέματα Θα ήθελα να σα ζητήσω στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις για τον Brexit που θα δούμε πώς θα ολοκληρωθούν να προσέξετε όχι μόνο το Γιβραλτάρ που οπωσδήποτε πρέπει να το προσέξετε αλλά και το θέμα των σαλίες και της αμοιβαία πρόσβασης σε νερά και πόρους. Πολλά συμφέροντα ευρωπαϊκά, ισπανικά και τις περιοχές μου της Γαλλικίας. Ε, ε, ε, θέλω να σας τονίσω ότι το νέο πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο και τα νομικά, νομοθετικά κύματα της Κομισιόν δεν αφήνουν σε καλή θέση τις περιφέρειες της Ισπανίας που μπορεί να υποστούν μεγάλες περικοπές. Παρακαλώ να το προσέξετε πάρα πολύ. Herr Präsident, ich freue Κύριε Πρωθυπουργέ, χαίρομαι που μας κάνατε σήμερα την τιμή να βρίσκεστε εδώ σήμερα. Ελπίζουμε σε εσά, ελπίζουμε ότι με το νέο ύφο σας στην πολιτική θα βοηθήσετε να προοδεύσει η Ισπανία. Αντί για αντιπαράθεση, ε, ε, στις διαπραγματεύσεις ε, έχετε εισάγει ένα πιο συνενετικό κλίμα και αντί για πολιτική λιτότητα ε, προσπαθείτε να δημιουργήσετε οικονομικά κίνητρα για οικονομική ανάπτυξη και ισορροπημένο προϋπολογισμό. Ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Όσον αφορά τα μέτρα στην αγορά εργασίας, ε, ανακαλείτε τα μέτρα της, ε, του προκατόχου σας που προσπάθησε να ε, περιορίσει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχει το λόγο ο κύριος Σάντσεθ για να απαντήσει ερωτήσει των Ευρωβουλευτών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ όλους τους Ευρωβουλευτές που αξιοποίησαν την ευκαιρία αγόρευσης. Και θα ήθελα να σας ε, ευχαριστήσω γιατί πραγματικά ε, αυτή η ένταση ζω, ζωγονεί την ε, συζήτηση. Υπήρξε μεγάλος αριθμός παρεμβάσεων διαφορετικού πολιτικού στίγματος. Εγώ θα προσπαθήσω να απαντήσω στο σύνολό τη όχι την καθεμία ξεχωριστά, βάσει των αξώνων, ε, των θεματολογικών αξώνων τους. Ε, και καταρχήν όσον αφορά τον, το πολυμερές ε, πνεύμα και τα όσα αναφέρθηκαν για τον φεντεραλισμό είπα ότι η κυβέρνηση ε, υπερασπίζεται την πολιτική ατζέντα πολιτικής αλλαγής. Πιστεύουμε ε, την ατζέντα 30 βάση του ενός, πολυμερούς, ενός πνεύματος πολυμερούς συνεργασίας και θεωρώ ότι συμφωνεί με τα όσα είπα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ισότητα των Φύλων και επίσης τα όσα κάνουμε στην Ισπανία, την έγκριση κάποιων μέτρων που αφορούν την, τον αγώνα κατά της ε, έμφυλης ε, βίας υπέρ της ισότητας των φύλων ή την έγκριση νόμων που μειώνουν το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στο εργασιακό περιβάλλον. Και θα ήθελα εδώ να προσθέσω κάτι. Ορισμένοι παρεμβαίνοντες μίλησαν για την ανεργία που είναι απαράδεκτη στην Ισπανία με σχετικούς ε, χώρους, αν συγκρίνουμε με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και όσον αφορά την ένταξη στην Ευρωζώνη. Αλλά επίση θα σας πω το εξή. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν... Ε, ε, είναι η πρώτη φορά όπου 48% ε, των όσων ε, είναι κοινωνικά ασφαλισμένοι ε, στην Ισπανία είναι γυναίκες. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Ισπανίας που οι γυναίκες έχουν ενταχθεί με τον τρόπο αυτό στην αγορά εργασίας. 22% έχουν ελάχιστες αποδοχές. Είναι πρώτη φορά στην ιστορία, στη δημοκρατική ιστορία της χώρας μας, όπου ένα πολύ μεγάλο ποσοστό γυναικών είναι καλυμμένοι από το ασφαλιστικό σύστημα. Άρα λοιπόν η ισότητα των φύλων, επίσης αγώνας κατά της ε, παιδικής φτώχεια. Εμείς ε, όχι μόνο θέσαμε την ανάγκη ενίσχυσης ε, της ε, εγγύησης για τα παιδιά, αλλά και, και σε επίπεδο ε, προσπαθούμε να πατάξουμε την παιδική φτώχεια ενισχύοντας όλα τα μέτρα που συνδέονται με την εγγύηση για τα παιδιά ε, προσπαθώντας να την μεταφέρουμε από το νοσιακό στο ισπανικό επίπεδο. Όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, ορισμένοι ομιλητές αναφέρθηκαν στο βαθμό δέσμευση τη ισπανική κυβέρνηση σε σχέση με το θέμα αυτό. Πρόκειται να εγκρίνουμε σύντομα ένα νόμο για την κλιματική αλλαγή, μια εθνική στρατηγική για την κλιματική μετάβαση, ε, ε, ούτως ώστε η μετάβαση αυτή να είναι δίκαιη ε, σε εκείνες τις βιομηχανικές ζώνες της Ισπανίας να βρεθούν κάποιες λύσεις εν σχέση με όσων πλήττονται. Επίση, ορισμένοι εμιλητές ε, αναφέρθηκαν σε ένα ευρύ πακέτο δικαιωμάτων και ελευθεριών ε, που εκπώνησε συντηρητική κυβέρνηση. Μιλήσατε για τον ε, νόμο Φήμετρο, για όλα όσα έχουν να κάνουν με την εργασιακή μεταρρύθμιση και τα διεργατικά δικαιώματα των εργαζομένων στη χώρα μας. Να σας πω τα εξή. Σε σχέση με τον νόμο φήματρο είναι τώρα σε διαδικασία τροποποίηση ε, και ελπίζω πως θα μπορέσει να εγκριθεί ε, από τον Φεβρουάριο και μετά. Και όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα, να σας πω ότι η κυβέρνησή μας ε, προωθεί το κοινωνικό διάλογο. Σε 7 μόνο μήνες έχουμε εγκρίνει ένα σχέδιο για την απασχόληση των νέων για να μειωθεί σε 3 χρόνια το ποσοστό των ε, νέων ανέργων κατά τρία ποσοστιαίες μονάδες. Επίσης έχουμε φτιάξει ένα σχέδιο αγώνα ε, καταπολέμησης μάλλον της επισφάλειας στην αγορά εργασίας ε, και έχουμε διαπιστώσει ε, και μετατρέψει μάλλον διάφορες μορφές συμβάσεων που ήταν παράνομες στην ουσία σε αορίστου χρόνου ε, συμβάσεις. Στη χώρα μας έχουμε 3, 3 ε, εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες που θα βρουν δουλειά, συμφωνία μεταξύ των συνδικάτων και των εργοδοτών με κάλυψη για τα εργατικά ατυχήματα και ούτω καθεξής. Άρα ε, λοιπόν ε, ε, πλεύρη προσπάθεια σε επίπεδο ισπανικό αλλά και σε επίπεδο ευρωπαϊκό και θέλω να κάνω δύο ε, επιπλέον ε, ε, σκέψεις που προέκυψαν σε σχέση με την εξωτερική πολιτική και τη σχέση με τη Βενεζουέλα να σας πω ότι η κυβέρνηση της Ισπανίας αλλά και ως αρχηγός αντιπολίτευσης προηγούμενα δεν αναγνωρίσαμε την νομιμότητα των εκλογών της χώρας αυτής ούτε αναγνωρίσαμε τον ε, Μαδούρο. Ε, η απόδειξη είναι ότι δεν ήμασταν παρόντες όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του. Έχουμε συστηματικά ζητήσει και επανελειμμένα από το καθεστώς του Μαδούρο να ελευθερώσει τους πολιτικούς κρατούμενους. Ε, χάρη στην καλή διαχείριση του Υπουργού Εξωτερικών καταφέραμε να μπορέσουν κάποιοι κρατούμενοι να έρθουν στην Ισπανία και είχα την ευκαιρία μάλιστα να μιλήσω μαζί τους και σίγουρα η θέση που έχει η κυβέρνηση της Ισπανίας ε, για το θέμα της Βενεζουέλας είναι να προσπαθήσουμε να, ε, να φτιάξουμε μια συμμαχία, ένα, μια ομάδα διευκόλυνσης του διαλόγου που θα αποτελείται από χώρες ευρωπαϊκές αλλά και από χώρες της ομάδας της Λίμα. Δεν συμμετείχαμε στην απόφαση που πρόθεσε η ομάδα της Λίμα και να σας πω ότι η κυβέρνηση της Ισπανίας δεν έχει την ίδια ίδια ιδέα. Προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ομάδα διευκόνησης που ακριβώς αυτό που κάνει είναι να επιτρέψει μια διέλευση με το, μια, ένα διάλογο ε, Επίση, θα πρέπει να μιλήσουμε για τη μεταναστευτική κρίση στη Βενεζουέλα. Ε, να πούμε ότι ε, είναι πολλοί οι Βενεζουαλάνοι που ζητούν άσυλο στη χώρα μας, αλλά επίσης η κρίση της μετανάστευσης ε, ε, στην Λατινική Αμερική, στην Κολομβία, Βραζιλία, Χιλή, με πολλές χώρες που μπόρεσα να συζητήσω αυτούς τους ε, μήνες που είμαι πρόεδρος της κυβέρνησης, να σας πω, ως το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ο υπουργό μα αλλά και η κυβέρνησή μα προσπάθησε να απεμπλέξει, να απελευθερώσει πόρου για να βοηθήσει τι χώρε αυτέ ώστε να διαχειριστούν με λογικό τρόπο την ε, εισρωή προσφύγων που αντιμετωπίζουν και ιδιαίτερα την Κολομβία που ε, ε, την οποία στηρίζουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Για τα Κανάρια νησιά, η κυβέρνησή μας ε, να σας πω ότι σε λίγο περισσότερο από 7 μήνες ξεκίνησε τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος των Καναρίων και υπέγραψε όλα τα συμβούλια. Δεν, κάνουμε, δεν φτιάχνουμε υπερπεριφερειακές περιοχές, ε, εμείς στηρίζουμε τα δικαιώματα των, ε, της περιοχής αυτής. Και να πω και κάτι γενικά, τέλος σε σχέση με τις ε, παρεμβάσεις του εκπροσώπων του ΕΛΚ ε, του Λαϊκού Κόμματος και το θέμα της Καταλωνίας. Το είπα και στην Ισπανία και θέλω να το πω και στους Ισπανούς Ευρωβουλευτές. Να σας πω ότι η μερίσια διάταξη της δεξιάς ε, σημαίνει μάλλον περισσότερο χαρακτηρίζεται από την ακροδεξιά σε δύο θέματα. Πρώτον, το να χρησιμοποιηθεί η Καταλωνία, δηλαδή η συνοχή και η συμβίωση, ως ένα στοιχείο για να κάνετε αντίσταση στην κυβέρνηση της Ισπανίας που θα είναι και θα είναι είναι και θα είναι η σοσιαλιστική κυβέρνηση και τηρεί το Σύνταγμα όσο είμαστε στην αντιπολίτευση και όσο είμαστε στην κυβέρνηση. Και θα ήθελα και το Λαϊκό Κόμμα να κάνει το ίδιο εφόσον είναι στην αντιπολίτευση. Δεύτερον, αν πρέπει να δω για να βρω κάποιο τρόπο διακυβέρνησης που αποσταθεροποιηθεί περιοχές και χώρες, περισσότερο είναι το το, το ελβετικό μοντέλο και παρά αυτό το οποίο είδαμε μόλις στην Ανδαλουσία. Eh, Σας ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε της Κυβέρνησης της Ισπανίας. Σας ευχαριστούμε που απαντήσατε στις ερωτήσεις των βουλευτών. Πιστεύω πως αυτή η συζήτηση ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έγινε πολλής λόγος για την Ισπανία, αλλά και για την Ευρώπη, ε, για την πολιτική της Βενεζουέλας για μας είναι κάτι σημαντικό. Εμείς πειρασπίζουμε το δικαιώματα των πολιτών της Βενεζουέλας. Δεν μπορούν να πεθαίνουν από την πείνα σε αυτή τη χώρα που δεν υπάρχει ούτε ελευθερία ούτε δημοκρατία. Ευχαριστώ όλους. Onorevole Viotti, chiede la parola? Sì. Καθίστε παρακαλώ. Ναι, μόνο ένα λεπτό να κλέψω από το χρόνο των ψηφοφοριών, γιατί Πολλές πηγές ε, δημοσιογραφικές λένε πως ε, στην Τσετσενία έχουν γίνει δεκάδες συλλήψεις ε, ενάντια σε ομοφιλόφιλους και τρεις νεκροί υπάρχουν μόνο και μόνο επειδή είναι ομοφιλόφιλοι. Δεν μπορούμε να είμαστε μόνο οικονομία και χρήματα. Στις σχέσεις με τη Ρωσία, εγώ ευχαριστώ την Επίτροπο Μογκερίνη γιατί του <coughs> θύμισε ε, στον Υπουργό. Δεν μπορούν οι σχέσεις μας με την Ρωσία να είναι μόνο οικονομικές. Είμαστε οι πρωταθλητές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να θυμίσουμε στην Ομοσπονδία ε, τη Ρωσική να, ανοίξει, ξεκινήσει έρευνε για το τι γίνεται στη Τσετσενία. Δεν μπορεί να δολοφονούνται άνθρωποι επειδή είναι ομοφιλόφιλοι τη σήμερον ημέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βιώτη. Στην έναρξη της συνεδρίασης της Δευτέρας 14 Ιανουαρίου ε, αναφέρθηκαν οι αποφάσεις διαφόρων επιτροπών να ξεκινήσουν διοργανικές πραγματεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 1. Ε, να θυμίσω ότι έλαβα έτοιμα από το ECR και από διάφορους βουλευτές να θέσουμε σε ψηφοφορία το αίτημα της Επιτροπής Γιούρη να ξεκινήσουν προματεύσεις σε σχέση με την έκθεση περί διασυνοριακών συγχωνεύσεων ή αποσχέσεων με τη συγκίτρια την κυρία Ρέγνερ. Έλαβα επίσης από πλευρά των Πρασίνων ε, και τη ΣΑΛΤΕ το αίτημα να, ψηφιστούν, να ψηφιστεί η απόφαση της Επιτροπής ΕΠΕΚ για έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων για τις εκθέσεις σε σχέση με το πολιετές πρόγραμμα για την αλληλεία για τα βενθοπελαγικά είδη στην Δυτική ε, Μεσόγειο. Κλάρα Εουτζένια, Βιέρα Γκαρσία είναι οι εισηγητέ. Οι ψηφοφορίε αυτέ θα γίνουν αύριο. Όσον αφορά τις άλλες αποφάσεις για έναρξη διαπραγματεύσεων διαθεσμικών που διαβιβάζονται αντίστοιχα στην Επιτροπή ΕΚΟΝ, στη και στην ΤΡΑΝΑ, δεν έχω λάβει κανένα αίτημα ψηφοφορίας. Αυτές οι επιτροπές λοιπόν μπορούν να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις. Ξεκινάμε με τις ψηφοφορίες. Πρώτη ψηφοφορία, κλείσιμο των λογαριασμών για την υπηρεσία υποστήριξη για το άσυλο για το οικονομικό έτος 16. 2016 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε σχέση με τις συμφωνίες Ένωσης Μαρόκου, ονομαστική κλίση, άρχεται. votazione è Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ευρωπαϊκή Ένωση Μαρόκο τροπολογία για την Ευρωπαϊκή Μεσογειακή Συνεργασία, παράγραφος 9, σε δύο τμήματα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τρία, υπέρ, κατά, αποχές. Θα το ελέγξουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, επαλήθευση ηλεκτρονική άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 1. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Με ονομαστική ψηφοφορία, το ψήφισμα στο σύνολό του, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Και τώρα θα έρθουμε και πάλι στην τροπολογία 1 και 4 για τη μεσογειακή συνεργασία, ονομαστική ψηφοφορία, Άρχιετη ψηφοφορία. Για την έκθεση ΣΑ και πάλι. Πέραση ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Κύριε Σεκόφσκι, θέλατε το λόγο, παρακαλώ. Θα ήθελα να, να θυμίσω σε όλους ότι είναι εδώ παρόντες ε, οι φίλοι μας από το Μαρόκο, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν να τους καλωσορίσω. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψή σας εδώ. Και τώρα θα έρθουμε στην έκθεση Winkler, Ευρωπαϊκή Ένωση Κίνα. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Έκθεση αρένα. Ε, μπορείτε να έχετε το λόγο για ένα λεπτό, αν το επιθυμείτε, κυρία Αρένα. Παρακαλώ, στο μικρόφωνο όμως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 έχει ως αντικείμενο να δοθεί η δυνατότητα στον κλάδο να υποστηριχτεί η οικονομία. Είναι σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στους εργαζόμενους. Επίσης είναι σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στους εργαζ... στις επιχειρήσεις για να υπάρξει συγκεκριμένη απόκριση στα προβλήματα απασχόλησης. Ε, αυτό είναι το περιεχόμενο της τροπολογίας 96 και επιθυμώ να έχω την υποστήριξή σας. Τώρα θα περάσουμε στην ε, τροπολογία, ε, στην, ε, συγγνώμη, στην ψηφοφορία. 1, 21, 23, 27, 29, 52. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 22 στη δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκ... απορρίπτεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 62 υπέρ, κατά. Αποχές, ε, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 62. Άρχεται η ψηφοφορία. Κιούσα. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 73. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 85. Υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται τέλος ε, να ήταν δύσκολο αλλά εγκρίνεται ε, τροπολογία 98 ονομαστική κλίση α, συγγνώμη 98 διορθώνει ο πρόεδρος, ε, με διανατάσσεω της χειρός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 96 ονομαστική κλίση, άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται. 97 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 28 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ε, ναι, απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Ψήφιση της πρότασης Επιτροπής με ονομαστική κλίση άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην εισηγητρία και θέλετε να παρέμβετε. Δεν θέλετε. Πρώτη ανάγνωση λοιπόν του Κοινοβουλίου έτσι ολοκληρώθηκε. Passiamo alla relazione για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Τροπολογίες 1 και συνέχεια. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 40. Ονομαστική κλίση άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται 97. Ονομαστική κλίση. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 171. Ονομαστική κλίση άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 89. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 168. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 89. Υπέρ. Κατά αποχές έγκρινεται 89 CP3 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές έγκρινεται 89 πάλι 4 υπέρ κατά αποχές απο, εγκρίνεται 172 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 89 cp 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 173 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 174 υπέρ α, συγγνώμη είναι ονομαστική κλίση 174 άρχεται τέλος απορρίπτεται 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 92 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική κλίση, άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. 162. Άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. 175. Ε, άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται. 92. Ποια είναι υπέρ. Κατά αποχές έγκρινεται. 176. D. Ονομαστική κλίση. Άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 177, ε, ε, ονομαστική κλίση, άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται. 92, πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική κλίση. Τέλος. Εγκρίνεται. 178 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 179 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 163 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 179 169 ε, με συγχωρείτε άρχεται πέρας απορρίπτεται 164 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 170 ε, ονομαστική κλίση άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 167 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 161 ονομαστική κλίση άρχεται πέρασε Απορρίφθηκε. Η ψηφοφορία της πρότασης της Επιτροπής, όπως τοποποιήθηκε, μονομαστική κλίση, άρχεται. Έρας, εγκρίνεται. Κύριε Λόπε Φοντανιά, θέλετε να πάρετε το λόγο, μπορείτε. Ευχαριστώ. πολύ κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνα με το κανόνα 524 ε, επιθυμώ η έκθεση να επανέλθει στην, ε, να αναπευθεί στην Επιτροπή. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Οπότε ψηφίζουμε την πρόταση της εισηγήτριας. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παραπέμπεται λοιπόν στην αρμόδια επιτροπή για την έναρξη των διοργανικών διαπραγματεύσεων. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Περνάμε στην έκθεση αρήμων, ειδικέ διατάξει που διέπουν το στόχο Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία. Τροπολογίε από το 1 μέχρι το 199. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχέ γίνεται. 101. Άρχεται. Συγγνώμη, 201 είπε, ε, άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται. Καταπίπτει η τροπολογία 200 και ψηφίζουμε την πρόταση της Επιτροπής με ονομαστική κλίση. Ποιος ζήτησε να παρέμβει? Όχι, όχι, μισό λεπτό. Είμαστε στη μέση της ε, ψηφοφορίας. Έχει αρχίσει η ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Τέλος. Εγκρίνεται. Αν θέλετε να παρέμβετε τώρα. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους συναδέρφους που συνέβαλαν ε, στην εκπόνηση του εγγράφου αυτού. Μετά από την χθεσινή ψηφοφορία για το Brexit στο Λονδίνο. Νομίζω ότι ε, είναι ε, αρκετά αισιόδοξα τα μηνύματα αυτά εδώ πέρα. Ε, το Interreg προβλέπει και την εδαφική συνοχή. Και επίσης προσλέπω στην έναρξη των διαπραγματεύσεων σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού. Ευχαριστούμε κύριε Αριμών, οπότε ψηφίζουμε για το σύνολο. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή για την έναρξη των διοργανικών διαπραγματεύσεων και φτάνουμε στην έκθεση Κβίσχου του Ροχόλτ για την ε, για την κατανομή των δεσμολογικών ποσοστώσεων περιλαμβάνοντας το πίνακα από έτη Ένωση και μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Ψηφίζουμε την τροπολογία 17. Υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 19. Υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ε, εγκρίνουμε το με τη 17 μάλλον ολοκληρώθηκε η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου και περνάμε στην έκθεση Λίνσες Stars, η Ενωσιακή Διαδικασία Έγκρισης Φυτοφαρμάκων της Ένωσης. Είναι η τελευταία έκθεση, αλλά είναι και η πιο μεγάλη. Έχουμε τις τροπολογίες 103. Άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 137. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 157 ε, ονομαστική κλίση άρχεται. Πέρας. Τροπολογία 56 είναι συγχωρείτε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 104. Ε, ονομαστική κλίση άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 105. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 57 δέλτα. Ψηφίζουμε. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. 106 ψηφίζουμε μονομαστική κλίση. Τέλος. Απορρίπτεται. 157, ε, συγγνώμη, 57 D, ε, άρχεται, πέρας, Απορρίπτεται. 58. Άρχεται. Τέλος. Καθαρά είναι. 59. Άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. 60. Άρχεται. πέρασε, Απορρίπτεται. 138. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 112. Ε, άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 61. Ε, άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 62, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Παράγραφος 12 του αρχικού κειμένου, άρχεται η ψηφοφορία. καλησπέρας. Γκρίνεται. Η 63 αν... ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε ψηφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 139. Καταπίπτει η 64. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 120. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 140. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 141. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 65. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 66. Ψηφίζουμε. η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 121. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 122. Ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. 123. Ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. 124 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 125 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 143 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 67. Ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. 144 υπέρ. Συγγνώμη. Αν ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. Η, 100, η 68 ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. Η 145 υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. 69 ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. Η 70 υπέρ. Έκλεισε. Απορρίπτεται. Η 71 ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. Η 72. Ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. Η 73. Ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. 75. Ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. 76. Ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. 77. Ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. Η 78. Ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα ψηφίζουμε. Έκλεισε. δεκτή. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Έκλεισε. Δεκτή. Τρίτο τμήμα Ψηφίζουμε. Έκλεισε. Δεκτή. Η 79. Ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. 80. Ψηφίζουμε. Έκλεισε. απορρίπτεται. Η 146 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 147 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 81 ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. Η 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 82 ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. Η 148 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 83 ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. 84 ψηφίζουμε. Έκλεισε. απορρίπτεται. 85. Ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. 133 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Ε, ε, δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Ε, επαλήθευση ψηφίζουμε.